έτσι ώστε να γίνονται ε, συγκεκριμένοι και δραστήριοι έλεγχοι της αγοράς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Ανακοινώνω ότι λάβαμε μία πρόταση ψηφίσματος. Η συζήτηση έκλεισε και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12 το μεσημέρι. Η επόμενη συνεδρίαση προβλέπεται αύριο 14 Ιουνίου από τις 9 στις 14 και 15 έως 17. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λύεται η συνεδρίαση και σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς.